Okay, dear colleagues, please take... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε. Second item. Δεύτερο σημείο της προτινόμενης ημερήσιας διάταξης είναι η έγκρισή της. Υπάρχουν επιθυμίες για τροποποίηση ή αλλαγή της ημερήσιας διάταξης. Εάν όχι, εγκρίνεται. Σημείο 3. Πρακτικά. Όπως συνηθίζεται, εάν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν υπάρχουν ενστάσεις ή αντιρρήσεις, τότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Έτσι λοιπόν θα γίνει. Σημείο 4. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη, όπως γνωρίζετε. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχετε πώς συμπεριφέρεστε και να προσέχετε τι λέτε. Την περασμένη εβδομάδα Μία αντιπροσωπεία μας πήγε στην ε, Νότια Κορέα και είχαμε θετικά αποτελέσματα σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, η οποία τώρα θα ισχύει για πέντε χρόνια. Και παρά τα προβλήματα που είχαμε με τη δική μου πτήση, πιστεύω πως η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή, όπως και η προετοιμασία. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε πολύ τη Γραμματεία, την ΧΕΙΚΗ τον Λέων Χεϊκή και τον Ματία. Άριστη λοιπόν η προετοιμασία της αποστολής. Συναντηθήκαμε με πολλούς ε, υψηλόβαθμους αξιωματούχους, με υπουργούς, με εκπροσώπους του εμπορικού κλάδου και συζητήσαμε την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, τον στον τομέα ICS αλλά και στην βιομηχανία. Συζητήσαμε επίσης το ενδεχόμενο μιας επιπλέον συμφωνίας πρόσθετης. Σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλή αποστολή και θα διαβάσετε τα σχετικά στην έκθεση. Τώρα, σχετικά με τη Μερκοσούρ. Συζητήθηκε το θέμα στην τελευταία ολομέλεια. Το θέμα της πρόσβασης στην αγορά. Ελπίζουμε λοιπόν να ενταθούν οι διαβουλεύσεις. Επίσης, στην τελευταία ολομέλεια είχαμε και το ψήφισμα για το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και ευχαριστώ όλους όσοι εργαστήκατε γι' αυτό. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά και να σας πω ότι αν και αναγνωρίστηκε στη Νέα, στην Νότια Κορέα το ψήφισμα, εμείς συζητήσαμε τις συνέπειες αυτού. Φιλιππίνες. Άρχισε ο πρώτος κύκλος συνομιλιών για μια μελλοντική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες. Ελπίζω να η πολιτική αλλαγή στις Φιλιππίνες να μην αλλάξει και την άποψη της κυβέρνησης για τη συμφωνία. Κανείς όμως δεν ξέρει ακόμα τις προθέσεις του νέου Προέδρου. Όπως γνωρίζετε, καμιά φορά οι απόψει του είναι κάπως προβληματικές σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θανατική ποινή κτλ. Σχετικά με την TIs. Το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα αυτό στην τελευταία συνεδρίαση των Υπουργών Εμπορίου Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Φαίνεται όμως μία τάση για συνέχεια στη συζήτηση. Και παρά το γεγονός ότι συζητήθηκε ο εξυγχρονισμός του, των ε, TDI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετήθηκε για τις ε, δικές της για τα δικά της αποτελέσματα των ε, ερευνών. Έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πόρισμα στην ιστοσελίδα της σχετικά με αυτό. Μπορείτε να το βρείτε για τα TDI. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω και θα περάσουμε τώρα μέσα στο σημείο 5. πληροφόρηση σχετικά με το, με το συνεχιζόμενο τριμερή διάλογο. Συζητήθηκε στον τελευταίο τριμερή διάλογο το θέμα των ορυκτών που προέρχονται από ε, εμπόλεμες περιοχές. Παρατηρήθηκε πνεύμα συνεργασίας, θέληση συμβιβαστική. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τα αποτελέσματα των συζητήσεων στην τελευταία του συνεδρίαση και θα συζητηθεί και στη συνέχεια με τους συναδέλφους από τα άλλα κράτη-μέλη στις 25 του μήνα, αυτή την εβδομάδα δηλαδή. και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα ορίσουμε και την ημερομηνία για τον επόμενο τριμερή διάλογο. Θα ήθελα όμως τώρα να δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Βίγκλερ, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω πολλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι η σχέση ανάμεσα στην Προεδρία και τα κράτη-μέλη είναι κάπως έντονες. Έχουμε κάποια σημάδια, κάποιες ενδείξεις από την Προεδρία, όμως δεν γνωρίζουμε αν έχουν και τα κράτη-μέλη παρόμοια θέση. Εδώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε δείξει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγάλη ευελιξία και πρέπει να καταστεί σαφές ότι υπάρχει ακόμα σημαντική απόσταση ανάμεσα σε αυτό που εμείς προσδοκούμε και σε αυτό που έχει προταθεί από το Συμβούλιο και την ετοιμότητα και τη διάθεση του Συμβουλίου να συζητήσει τις ε, φιλοδοξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν τρία κύρια θέματα τα οποία είναι ακόμα προς ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ε, downstream εφοδιαστικής αλυσίδας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να παρετηθεί των ε, ετοιμάτων του. Επίσης, συζητήθηκαν οι τεχνικές πτυχές της αναγνώρισης και η αναθεώρηση του κανονισμού. Είναι ακόμα υποσυζήτηση όλα αυτά. Οι πολιτικές ομάδες πιστεύω είχαν μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Η διαπραγματευτική ομάδα έδειξε ενότητα. Είχαμε μια ενιαία θέση απέναντι από το Συμβούλιο και πιστεύω πως είναι ε, καλό να συνεχίσουμε με αυτήν την έννοια ενωμένη στάση. Πιστεύω πως σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν σε τεχνικό επίπεδο, όμως οι συνάδελφοι που συμμετείχαν σε αυτές τις συνεδριάσεις τεχνικού τύπου αναγνωρίζουν ότι είναι ένας πολύ περίπλοκος κανονισμός. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε τον τελικό μας στόχο. Ο τελικό στόχος του Κοινοβουλίου είναι να υπάρχουν αποτελέσματα. Αποτελέσματα που θα αλλάξουν τις ζωές των πολιτών, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τις συγκρούσεις στις περιοχές αυτές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκλερ. Δεύτερος ε, τριμερής διάλογος εν εξελίξη. για τον ε, κανονισμό κατά των βασανισμών. Είναι λίγο απογοητευτικά τα αποτελέσματα στο θέμα αυτό, γιατί το Συμβούλιο δεν είναι ε, σε θέση να υποβάλει κάποια σημεία προς διαπραγμάτευση. Γι' αυτό και ε, δηλώσαμε σαφώς ότι μόνο εάν το Συμβούλιο υποβάλει ένα επιπλέον συμβιβαστικό κείμενο, θα γίνει ένας επόμενος τριμερής διάλογος και επομένως το Συμβούλιο επέβαλε στη συνέχεια συμβιβαστικές προτάσεις και έχουμε προγραμματίσει έναν τριμερή διάλογο για αύριο το απόγευμα. Να δούμε λοιπόν ε, τι συμβαίνει. Δυστυχώς ε, η εισηγήτρια, η κυρία Τσάκ, δεν θα μπορέσει να είναι εδώ σήμερα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, είναι σε θέση να την ε, αντικαταστήσει. Όχι. Ευχαριστώ. Α, ο κύριος Τάκουλα. Μάλιστα. Δεν το ξέρε. Συγγνώμη. Λοιπόν, για το Ιράν. Όχι. Να αντικαταστήσετε την εισηγήτρια για να μας πείτε τα του τριμερούς διαλόγου. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο από την ομάδα σας, κάτι να πείτε. Ναι, εγώ έτσι ξέρω. Άμα πάμε στο 7 έχω να σας πω. Εντάξει, θα τα πείτε στο 7. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Συζητήσαμε αρκετό καιρό την ε, πολιτική εμπορίου για τον 21ο αιώνα και θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε την ανακοίνωσή της πέρσι και πλέον επαφείται σε μας να ε, δούμε μια πιο μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Έχουμε ορίσει την ησυχήτριά μας, η οποία μας ε, υπέβαλε την έκθεσή της και έχουμε και πάρα πολλές τροπολογίες. 414 στο σύνολο. Επομένως έχουμε πολλή δουλειά για τις επόμενες ε, εβδομάδες και μήνες αλλά βέβαια καθήκον ε, για να ε, παρουσιάσει την ε, έκθεση έχει η συγκητρία η κυρία Μπεγκίν και στην οποία θα δώσω και το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους και τις συγκητές για τα όσα έκαναν και για τη διάθεση που έδειξαν στην προηγούμενη συνεδρίαση στο Στρασβούργο να συμβιβαστούμε η εργασία μας για τις συμβιβαστικές ε, προτάσεις ε, προχωρά. Το πρώτο σχέδιο έκθεσης ε, έτυχε καλή υποδοχές από τους αδέλφους και τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και τώρα με τους του εισηγητές προσπαθούμε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις οι οποίες κατά την άποψή μου είναι σημαντικές. Όπως πολύ σωστά έλεγε και ο Πρόεδρος και όπως υπενθυμίζει και ο τίτλο, πρόκειται για μια στρατηγική για το μέλλον. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε ένα ε, κείμενο στραμμένο προς το μέλλον, αλλά και να δώσουμε και την ευκαιρία στην, ε, ε, να διευκρινίσουμε τις προτεραιότητές μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας σαφή μηνύματα, τα οποία θα είναι σταθερά και για την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, αλλά και για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και σήμερα ότι δεν είναι χρήσιμο να επικεντρωθούμε σε θέματα τα οποία έχουν ήδη καλυφθεί, και στα οποία έχει εκφράσει σαφέστατα το Κοινοβούλιο την άποψή του και για την TTIP και για την TISA και κατά την άποψή μου δεν θα χρειάζεται, να επαναλαμβάνουμε συνεχώς αυτά τα θέματα. Πρώτον γιατί θα μπορούσαν να απολώσουν τη συζήτηση και να είναι κατά της ε, ε, πλειοψηφίας η οποία θέλουμε να είναι και συνεκτική και δεύτερον γιατί υπάρχουν και αρκετά κείμενα τα οποία ε, θα αφορούν τα θέματα αυτά και θα γίνουν ε, δεκτά. Θα ήθελα λοιπόν να μην επαναλάβουμε στις εργασίες μας αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί στο παρελθόν, αλλά να έχουμε ένα νέο κείμενο, σαφές, ξεκάθαρο, το οποίο θα καθορίζει κάποιες προτεραιότητες. Ελπίζω να μπορέσουμε να εργαστούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, με την ίδια θετική προσέγγιση που υπέδειξαν οι συνάδελφοι και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και να επενθυμίσω στους κοιόδης ηγητές ότι αύριο το απόγευμα 6.30 με 8 θα συναντηθούμε για να συζητήσουμε τις επόμενες συμβαστικέ προτάσεις οι οποίες έχουν ήδη διανεμηθεί ε, σήμερα μετά το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Κάσπαρη απουσιάζει. Υπάρχει κάποιος που τον αντικαθιστά στη σημερινή συνεδρίαση. Όχι. David Μάρτιν λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Τιτσιάνα για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της ότι όντως σημειώνουμε πρόοδο στις συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών. Το είχαμε πει και στο παρελθόν, το ξαναλέω και τώρα, ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το σχέδιο έκθεσης Υποβάλαμε εμεί 76 τροπολογίε παρόλα αυτά και το κάναμε προκειμένου να αποσαφηνίσουμε κάποια σημεία τα οποία δεν ήταν ξεκάθαρα, τα οποία απουσίαζαν από το αρχικό κείμενο. Ω σοσιαλιστέ, θέλουμε να τονίσουμε ότι ε, λέγεται αυτό στον βαθμό στο κείμενο. Πάντως είναι σημαντικό να πούμε ότι οι διευθετήσει ε, για τι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου θα πρέπει να αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη λύση. Πρέπει να προωθήσουμε το πολυμερέ εμπορικό σύστημα. Το επαναλαμβάνουμε αυτό και πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του πολυμερού συστήματος δεν καταφέρουν να σημειώσουμε την ευκταία πρόοδο. Επίσης, κατά δεύτερο λόγο, το έχουμε πει και σε άλλη έκθεση αυτό, δεν θέλουμε απλώς κεφάλαια όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία είναι καθαρά συμβολευτικά, αλλά θέλουμε τα κεφάλαια αυτά να είναι εφαρμόσιμα, να μπορούν να επιβληθούν στα πλαίσια των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Νομίζω ότι επίση δεν θα πρέπει να συμφωνούμε απλώς για νέες συμφωνίες και συνθήκες, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται και στην πράξη. Στην αποστολή που είχαμε στην Κορέα την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχουμε τη σωστή εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Θέλουμε ένα υψηλότερο βαθμό διαφάνειας και θέλουμε όσον αφορά το TTIP να έχουμε κάποια στοιχεία διαφάνειας τα οποία θα υπάρχουν και σε άλλες συμφωνίες Λαμβάντας υπόψη τη φύση του εμπορίου σήμερα, καθώς επίσης και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής να λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να ισχύουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, να μην περιορίζονται μόνο στην εδαφική επικράτεια της Ευρώπης, αλλά να καλύπτουν εδαφικά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης, θεωρήσαμε ότι κάποια στοιχεία υποεκπροσωπούνται κάπως στο κείμενο αυτό και έχουν να κάνουν με στοιχεία τα οποία έχουμε δει στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, το πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε τα μέσα εμπορικής άμυνας ή το πώς μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το ζήτημα του καθεστώτος οικονομίας αγοράς της Κίνας. Ξέρετε επίση ότι στο κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γίνεται καμία αναφορά στην περίοδο μετά την Κοτονού. Παρ' όλα αυτά, τονίζω ότι σημειώνουμε πολύ καλή πρόοδο, έδειξε ιδιαίτερη ευελιξία η εισηγήτρια. Καταφέρνουμε να πετύχουμε αυτή τη στιγμή ένα υψηλό βαθμό συνένεση και είναι πολύ σημαντικό, όπω είπε και η εισηγήτρια, να καταφέρουμε μέσω του εγγράφου αυτού να δώσουμε μια, ένα σαφή προσανατολισμό στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η αίμα τώρα έχει το λόγο. And... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζουμε να δείχνουμε αυτή τη στιγμή πόσο εμπλεκόμαστε στην εμπορική πολιτική από τον σημαντικό αυτό αριθμό τροπολογιών που έχουν ε, υποβληθεί. Θα μπορούσα εγώ να φωτίσω λίγο πιο θετικά τα πράγματα, να αναφερθούμε λίγο στις θετικές επιπτώσεις του εμπορίου, το πώς συμβάλλει στο να μειωθεί για παράδειγμα η φτώχεια. Γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια τροπολογιών μου, προσπαθώ να αναγνωρίσω ακριβώς αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, συμφωνίες διευκόλυνσης του εμπορίου, κυρίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες δυσκολεύονται πάρα πολύ να καταφέρουν να συμμορφωθούν γρήγορα με κάποιες πολύ πολύπλοκες τελωνιακές διαδικασίες. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να εναρμονίσουμε, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες αυτές προκειμένου από χώρες να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτές τις συμφωνίες διευκόλυνσης του εμπορίου και προκειμένου συμφωνίε αυτέ να μπορούν να έχουν επωφελεί τελικά επιπτώσει στι χώρε αυτέ, μειώνοντα συγκεκριμένα τα επίπεδα φτώχεια. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δραματίσει ένα πολύ σημαντικό θετικό ρόλο να βοηθήσει στο να ολοκληρωθούν και να οριστικοποιηθούν κάποιε εμπορικέ συμφωνίε, ιδίω αυτή που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή με τη Σιγκαπούρη αλλά και με τον Καναδά. Εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όντως συμβάλλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ολοκλήρωση των συμφωνιών αυτών, έχοντας κατά νου βέβαια το συμφέρον των πολιτών και των καταναλωτών. Μόνο αν οριστικοποιήσουμε γρήγορα τι συμφωνίε αυτέ θα καταφέρουν να συνειδητοποιήσουν οι πολίτε πόσο θετικέ είναι οι επιπτώσει αυτών των συμφωνιών. Το είπα και σε προηγούμενη συνεδρίαση, το λέω και τώρα, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ψηφιακή οικονομία καθώ επίση και στο μέλλον τη εμπορική πολιτική, ιδίω στα πλαίσια του cloud computing και άλλων τεχνολογιών, τεχνολογικών εξελίξεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των συμφωνιών αυτών να μπορούμε να ευθυγραμμιζόμαστε περισσότερο με τις νέες τάσεις που επικρατούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να ταινίσουμε περισσότερο το μέλλον όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές. Να ευχαριστήσω και εγώ πάντως την συγγήτρια. Στην έκθεσή της αναφέρθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο τους ε, στο σημερινό εμπορικό παγκόσμιο σύστημα. Στις δικέ μου τροπολογίε προσπαθώ να ενισχύσω τη διατύπωση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για το πώς θα μπορούσαν αυτές να σωματωθούν περισσότερο στην ε, παγκόσμια λυσίδα αξιών και πώς μπορούν να τα βγάλουν πέρα ιδίω όταν πρέπει να συμμορφωθούν με τι διαδικασίε αντι αντι-dumping. και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σημείο επαφή και εξυπηρέτηση όσον αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ιδίω όσον αφορά το TTIP. Αυτή είναι η τελευταία τροπολογία την οποία θα ήθελα να παρουσιάσω προς τους συναδέλφους την 388 όσον αφορά το παράνομο εμπόριο, την παράνομη λαθροθυρία και το πώς ουσιαστικά το φαινόμενο αυτό ζημιώνει πάρα πολύ σημαντικά τη βιοπικιλότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνει μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στο ζήτημα αυτό και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην έκθεση την οποία συντάζω αυτή τη στιγμή όσον αφορά την καταπολέμηση της λεφροφυρίας και τις δεινές επιπτώσεις που έχει για την βιοπικιλότητα. Προσβλέπω πάντως την αυριανή συζήτηση που θα έχουμε μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και με σίγουρο θα καταλήξουμε σε πιο θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Στάκουλα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρου ε, του σκιωδού εισηγητή των ε, Φιλελευθέρων. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίαση τη ε, υφιστάμενη κατάσταση. Όπως αναφέρθηκε η πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών έγινε πριν από δύο εβδομάδες και συζητήσαμε συμβιβαστικές προτάσεις. Πιστεύω πως ε, μπορώ να στηρίξω αρκετές από τις συμβιβαστικές προτάσεις, οι οποίες κιόλας συμπεριλαμβάνουν και τη δική μας θέση σχετικά με την εμπορική και επενδυτική πολιτική. Υπάρχει μια παράγραφος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να αναλάβουν ε, κατά τη ε, διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων. Πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να είναι μία από τις κυριότερες προτεραιότητές μας και πρέπει να φαίνεται σαφώς στην έκθεση. Επίσης, θα ήθελα να φαίνεται περισσότερο και η πρόθεση της ψηφιακής διάστασης του διεθνούς εμπορίου στην έκθεση. Η διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι ώστε να μπορούμε να συμμορφωθούμε με ε, τις ε, προδιαγραφές αυτής της τόσο φιλόδοξης ε, πρότασης. Σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας, πιστεύω πως χρειάζεται να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω πως υπάρχει ανάγκη να αναφερθεί στην έκθεση το θέμα της αποτελεσματικότητας των μέσων εμπορικής άμυνας Και τέλος θα ήθελα να πω πως όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2015 είναι ένα πολύ σημαντικό ε, τμήμα της ε, συμφωνίας TTIP. Είναι μια ε, συμφωνία με πολιτική βαρύτητα και η έκθεση πρέπει να συνδέεται με αυτό και να την στηρίζει σαφέστατα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ να συνεχίσω τις ε, διαβουλεύσεις για αυτή την τόσο σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για αυτές τις επικοδομητικές προτάσεις. Θα περίμενε κανείς να υπήρχαν πολύ περισσότερες τροπολογίες από τις 600 περίπου που υποβλήθηκαν. Διότι όσο πολλές είναι οι τροπολογίες, τόσο φαίνεται και πόσο πολύπλοκο θέμα είναι οι εμπορικές ε, σχέσεις. Στο Στρασβούργο φτάσαμε σε έναν πρώτο συμβιβασμό και πιστεύω πως ε, τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτά που προσδοκούμε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους σε πολλά που αναφέραν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, την δημοσίευση της εντολής. Αυτό πιστεύω πως είναι προαπαιτούμενο, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, πιστεύω πως πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στην ε, πολιτική ως μέσο και στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο στις τρίτες χώρες. Εδώ πιστεύω πως δεν επιτυγχάνεται ισορροπία και αυτό μπορεί να οδηγήσει πολύ γρήγορα στις αντίθετες εξελίξεις η συγγήτρια και εγώ ήμασταν μέλη της ε, αντιπροσωπείας ε, σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και συζητήσαμε στην τελευταία μας ε, συνάντηση θέματα, τα θέματα αυτά, το θέμα της, του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και οι συζητήσεις με τους Κινέζους εταίρους μας ήταν εξίσου δύσκολες. Μας εστάλει ένα σαφές μήνυμα ότι αν εσείς δεν μπορείτε να ε, αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της οικονομίας σας, αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Δεν φτάμε εμείς γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν περάσαμε έξι μήνες εντονότατων διαπραγματεύσεων με την ε, Κίνα και πιστεύω πως πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό. Πρέπει να σκεφτούμε ποιος μπορεί να είναι αυτός και σίγουρα συμφωνώ πως πρέπει να ζητήσουμε τον εξυγχρονισμό των ε, μέσων εμπορικής άμυνας με όλους τους εταίρους. Και φυσικά με την Κίνα. Έπειτα, όσον αφορά το fair trade, με χαροποιεί η αναφορά σε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούμε να το συνδυάσουμε και με το πρώτο σημείο και με την έλλειψη δηλαδή φιλοδοξίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα για ε, την κλωστοϊφαντουργία. Όταν αναφερθούμε στην κλωστοϊφαντουργία μπορούμε να ζητήσουμε βελτίωση της ε, στρατηγικής της Ένωσης. Και αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε με το πού θέλουμε να φτάσουμε στις πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες μας. Υπάρχει μια αναφορά στο σχέδιο έκθεσης, έχει συζητηθεί το θέμα στις διαβουλεύσεις, υπάρχουν και αποφάσεις του ΠΟΕ και πιστεύω πως ε, θα ήταν καλό να τις συνδυάσουμε. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα, στην ε, έμφυλη διάσταση της εμπορικής πολιτικής. Έχουμε τρεις γυναίκες στην Επιτροπή μας από διάφορες πολιτικές ομάδες οι οποίες προσπαθούν να ισορροπήσουν την ε, κατάσταση. Πιστεύω πως μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση εδώ και να υπάρχει μια αναφορά στην κοινή θέση του, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρχεντίνη. Εγώ δεν θα πατήσω σε αυτή την παρατήρηση ως γυναίκα, γιατί τελικά χρειάζεται να πρέπει να προστατεύεται ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην σας αφορά και απόλυτα. Λοιπόν, ε, για τα σχόλια που είπαν ο Ντέιβιτ Μάρτιν και ο Μάρτιν Σούλτς, οι πράσινοι προτιμούν πολυμερείς ε, εμπορικές συμφωνίες και έχουν πολλές επιφυλάξεις για τις διμερείς συμφωνίες. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα πρέπει ε, να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Όσον αφορά το εμπόριο και την ανάπτυξη. Υπάρχουν δύο στόχοι. Το να μην κάνουμε κακό και το να κάνουμε καλό. Πολύ συχνά δεν ε, ασχολούμαστε καν με το δεν κάνουμε κακό όσον αφορά την πολιτική εμπορίου για τις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλό δε μάλλον για το να κάνουμε κάτι καλό. Ε, όλα αυτά τα βλέπουμε στη συζήτηση για την TTIP, συζητούμε για το κατά πόσον θα έχουμε μισό της εκατό οικονομικής ανάπτυξης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα έπρεπε να συζητούμε τι θα σημαίνει αυτό για τις αναπτυσσόμενες χώρες και δεν αγγίζουμε καν το θέμα του ε, δεν προκαλούμε καμία ζημία, δεν κάνουμε κανένα κακό. Αναφέρθηκε και το ε, υπεύθυνο και δεοντολογικό ηθικό εμπόριο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, τα είδαμε και πριν από μία ώρα στην Επιτροπή Ανάπτυξης για τη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω της δέουσας επιμέλειας και στο κείμενό μας. Ε, θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναφέρουμε στο κείμενο. Υπάρχει και η σχετική τροπολογία 169 όσον αφορά το βιώσιμο εμπόριο και στο να μπορέσουμε να κάνουμε το καλό πιστεύουμε ότι χρειάζεται απαραίτητα δέουσα επιμέλεια υποχρεωτικά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ε, θα είμαι παρούσα στην ε, διαπραγμάτευση για τις συμβαστικές προτάσεις αύριο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέντινγκ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερο την εισηγήτρια για ένα πολύ καλό σχέδιο έκθεσης. Υπέβαλα κάποιες τροπολογίες οι οποίες επικεντρώνονται στα θέματα τα οποία με απασχολούν, τα γνωρίζει όλος ο κόσμος, ε, ε, η ψηφιακή τεχνολογία, η τίζα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φυσικά. Και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρεις από τις τροπολογίες, οι οποίες κατά την άποψή μου περιλαμβάνουν και την βασική στρατηγική και τη μεγαλύτερη πρόκληση για το μέλλον. Πρώτον, γιατί διαπραγματευόμαστε εμπορικέ συμφωνίες. Γιατί ε, χρειαζόμαστε σταθερούς ε, κανόνες του παιχνιδιού. Δεν πρόκειται πλέον για εμπορικούς κανόνες, αλλά για ένα γεωπολιτικό παιχνίδι και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Και δεύτερον, ποια είναι η εμπορική πολιτική που θέλουμε. Η άποψή μου είναι ότι ενισχύεται καθημερινά μία πολιτική ε, η οποία θα βασίζεται στην αμοιβαιότητα, με ισότιμο άνοιγμα από πλευράς αγορών, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να κρατήσει ορθάνυχτες τις πόρτες της και να δεχόμαστε να έχουμε εταίρους που θα τις έχουν ερμητικά κλειστές τις πόρτες τους. Επομένως, πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο μας και να διευκρινίσουμε σαφέστατα τα πράγματα. Και τρίτον, πώς διαπραγματευόμαστε. Και εδώ έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και για μένα το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ευθύ εξ αρχές μία σταθερότατη εντολή με κόκκινες γραμμές ε, οι οποίες θα έχουν αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρχει και μία ισχύς ε, για τους διαπραγματευτές μας ε, ενώπιον της οποιασδήποτε πρόκλησης. Είτε πρόκειται για διμερή πρόκληση, εγώ αντίθετα με τη συνάδελφο δεν είμαι αντίθετη σε διμερείς συμφωνίες, γιατί οι πολυμερείς συμφωνίες ξέρουμε ότι όλο ένα και περισσότερο δυσκολεύουν και επομένως αυτή η ισχυρή διαπραγματευτική εντολή είναι πάρα πολύ σημαντική για να μην χανόμαστε μετά σε ατέρμονες και άχρηστες συζητήσεις και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τη ε, διαπραγματευτική ικανότητα των διαπραγματευτών. Είδαμε τους ε, τελευταίους μήνες ότι αρχίζει να φουσά ένας νέος ε, άνεμος στις εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς την ουσία και ως προς τον, ε, τη μορφή και θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε αυτές τις αλλαγές. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγγήτρια έχει κάνει εξαιρετική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια, η Μακουλάδα, έχει το λόγο. Ε, θέλουμε και εμείς να συνεισφέρουμε ώστε να έχουμε την πληρέστατη και καλύτερη δυνατή έκθεση. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ε, πτυχές. Ε, νομίζω ότι όλα όσα είπε ο συντονιστής μας, ο Ντέιβιτ Μάρτιν και όλες οι τροπολογίες που έχουμε υποβάλει ως ομάδα και ε, όλα όσα θα κάνει ο Σκιώδης εισηγητής μας καλύπτουν πλήρως τις προτεραιότητές μας. Θα σταθώ λοιπόν σε τέσσερα πολύ συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, η ανάγκη να μεταρρυθμίσουμε την ε, πτυχή του φίλου στην ε, έκθεση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλάμε για την εμπορική πολιτική του μέλλοντος και να μην λαμβάνουμε υπόψη την ανάγκη να χρησιμοποιούμε το εμπόριο ως ένα μέσο για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων σε όλο τον κόσμο. Και επίσης πρέπει να εγγυηθούμε ότι η ισότητα των φύλων θα ε, είναι οριζόντια. Θα συμπεριλαμβάνεται δηλαδή με οριζόντιο τρόπο. Επίσης πρέπει να εγγυηθούμε ότι όχι μόνο θα συμπεριληφθεί ως απαραίτητο εργαλείο και ως κάτι το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να παρακολουθήσουμε κατά πόσον τηρούνται όλα όσα έχουν καλυφθεί. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο σε σχέση με το φύλλο. Δεν μπορεί να είναι τόσο καθυστερημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να υπογράφουμε καλέ συμφωνίε αν δεν έχουμε μέσα κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση. Γι' αυτό ακριβώ και ζητώ από την εισηγήτρια να υποστηρίξει την ε, τροπολογία 143. Δεύτερον, όπως σας έλεγα, δεν χρησιμεύει σε τίποτα να έχουμε καλές συμφωνίες εάν δεν συνοδεύονται και από την κατάλληλη εφαρμογή και να έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσουμε να δούμε πώς ε, μπορούμε να καλύψουμε όλες τις εργασιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και πώς επηρεάζουν αυτές οι εμπορικές ε, συμφωνίες και πώς καταφέρνουν να δημιουργήσουν ε, θέση απασχόλησης και ανάπτυξη, να βελτιώσουν την ευημερία των πολιτών και να βελτιώσουν και την ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό και ακριβώς πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένου δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί μπορεί να καταρτίζει μια ετήσια έκθεση, την οποία θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο, επί τη βάση αυτών των αξιολογήσεων. Χρειαζόμαστε ε, να μπορούμε να ε, διαβιβάσουμε στους πολίτες ε, τι εμπορική πολιτική υλοποιούμε, τι συνέπειες έχει και τι θετικά στοιχεία έχει. Και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ζητήσω και από την εισηγήτρια να υποστηρίξει την τροπολογία 194. Τρίτον, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί και αναθεώρηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί ε, να ε, είναι υποφελής για όλους όλες οι εμπορικές συμφωνίες και νομίζω ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρέπει να μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την πρόκληση που δημιουργεί το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων. Γιατί ορισμένες φορές μπορεί να είναι υποφελής οι συμφωνίες για τις επιχειρήσεις αλλά όχι για τους εργαζομένους. Γι' αυτό ακριβώς και θεωρούμε ότι θα πρέπει να μειωθεί το κατώτατο όριο πρόσβαση στο Ταμείο ώστε να μπορεί να είναι προ όφελο και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εργαζομένων αυτών των επιχειρήσεων, που είναι αυτέ που πλήττονται περισσότερο από τι συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό υποβάλαμε και την 409 τροπολογία. Και τέλο, θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια να δεχτεί την τροπολογία 260, την οποία υπέβαλα με στόχο να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική. Πιο συγκεκριμένα, την ανάγκη να έχουμε αίσιο τέλος το συντομότερο δυνατόν στη Συμφωνία για τη Μερκοσούρ και την ανανέωση των εμπορικών συμφωνιών με τη Χίλη και το Μεξικό. Συμφωνώ απόλυτα ότι ο σκιώδης εισηγητές μας και η εισηγήτρια θα μπορέσουν να καταλήξουν στους κατάλληλους συμβιβασμούς και ζητώ να λάβετε υπόψη τις τροπολογίες που υπέβαλα. Ευχαριστούμε κυρία Τεσσαρνές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω και εγώ δύο-τρία σημεία. Όντως η έκθεση αυτή ασχολείται με πολύ σημαντικά ζητήματα Πρώτον, λοιπόν, θεωρώ ότι το εμπόριο δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτό σκοπό. Πολύ καλό πράγμα το εμπόριο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί απότερο στόχο μας. Είναι απλώς ένα μέσο και αναφέρομαι αυτή τη στιγμή περισσότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να δούμε και τη δική τους την αυτάρκεια και πώς μπορούμε να την αυξήσουμε και όχι μόνο να προωθούμε τις εμπορικές σχέσεις με αυτές. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει επίσης και μια συνεκτικότητα με όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την εμπορική πολιτική. Και εδώ έχουμε πρόβλημα, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε κατακαιρματισμένα τις διάφορες πολιτικές χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους μια συνεκτικότητα. Τρίτον, χρειαζόμαστε διαφάνεια. Αυτό είναι ένα όρο εκ των ΟΥΚ άνευ, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε δημοκρατικέ συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γίνεται όλο και πιο σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πολλέ φορέ δεν υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια. Προχωρώ τώρα κάπω γρήγορα. Πρέπει όντω να έχουμε πολλέ μελέτε αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εξολογήσει αυτέ θα πρέπει όμω να είναι πιο διαφανεί, πιο συγκεκριμένε, καλύτερα εκπονημένες και νομίζω επίση ότι για κάποια ευαίσθητα προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε μνήε. Όπω μνήε οι συμφωνίε αυτέ θα πρέπει να υπάρχουν και σε ευαίσθητου τομεί, όπω ο υγειοργικό τομέα, ή για παράδειγμα ο οπτικοακουστικό τομέα, ή γενικότερα ο πολιτιστικό τομέα. Τομεί οι οποίοι δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου και επίση θα υποβάλω και τροπολογίε για όλα αυτά τα σημεία και όπω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, το λέω και εγώ, θέλουμε να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τα μέσα εμπορική μα άμυνα. Αυτό γίνεται πλέον επίγουσα ανάγκη. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την σημερινή συζήτηση θα ήθελα να τονίσω και εγώ ένα πράγμα εκ μέρους της ομάδας μου. Το εμπόριο με ξεκάθαρους και σαφείς κανόνες είναι φυσικά καλό είναι καλό και για τα καταστήματα, είναι καλό και για τους καταναλωτές και ε, για τους ε, εργαζόμενους, αν το δούμε παγκόσμια. Αν δούμε τι γίνεται τώρα στην Αφρική και την Ασία, παρατηρούμε ότι όποιος συμμορφώνεται με τους ε, κανόνες, τότε οδηγείται και στην ευημερία και, στην, ε, και στις καλές συνθήκες διαβίωσης. Αυτά φυσικά έχουν άμεση σχέση και εμείς ως ΕΛΚ υποστηρίζουμε την ε, αναφορά, την έντονη αναφορά σε αυτό, όπως έχει κάνει η, η συγγήτρια. Πιστεύω πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε, όμως θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ε, ταχύτατη στις ε, διαπραγματεύσεις, να γίνουν μεταφράσεις όσο το δυνατόν ε, συντομότερα και ε, με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις, έτσι ώστε να προχωρήσει η έκθεση για να οδηγηθούμε στην ε, συμφωνία. Ζητούμε λοιπόν την ε, γρήγορη ολοκλήρωση και των διαπραγματεύσεων και κύρωση της συμφωνίας για τους λόγους αυτούς. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρονται για την εμπορική πολιτική, για το εμπόριο αυτό, έχει φανεί πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια και πιστεύω πως τους οφείλουμε ε, μια σωστή και πλήρη ενημέρωση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να δώσουμε έναν πιο ανοιχτό χαρακτήρα στην ε, συζήτηση το άνοιγμα των ε, αγορών, για την ε, απελευθέρωση του εμπορίου, για τις ιδιωτικοποιήσεις κτλ. Πιστεύω πως ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να παραμερίσουμε τα εμπόδια που έχουν δημιουργήσει άλλες προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως και παράδειγμα η συμφωνία TPP που έχουν υπογράψει οι ΗΠΑ με τις χώρες του ελληνικού που είναι σίγουρα ε, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την δική μας βιομηχανία, ιδιαίτερα την αυτοκινητοβιομηχανία, όταν οι καταναλωτές της ΗΠΑ στρέφονται προς τις ιαπωνικές αγορές αντί για τις ευρωπαϊκές. Αυτό πιστεύω πως αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο για την βιομηχανία μας, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε. Η εισηγήτρια πιστεύω πως έχει συγγράψει ένα πολύ καλό σχέδιο έκθεσης, αρκετά ισορροπημένο. Πράγματι υπάρχουν εκατοντάδες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, αλλά πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα καταλήξουμε σε αρκετές συμβιβαστικές λύσεις. Πιστεύω πως πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ε, σύντομοι και περιεκτικοί και να μην χαθούμε στις λεπτομέρειες, αλλά να εστιάσουμε στην ουσία του πράγματος. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ακολουθήσουμε τις ε, προτάσεις και τη γραμμή της εισηγήτριας, διότι όπως σας είπα είναι μια αρκετά ισορροπημένη έκθεση και οι συμβαστικές ε, τροπολογίες πιστεύω πως ε, δεν θα είναι κάτι δύσκολο και σίγουρα δεν πρέπει να αποδυναμώσουν το μήνυμα και την ουσία της έκθεσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και προσβλέπω στις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Ο Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συνεχίσω κάτι που ανέφερε ο Ντάνιελ. Πιστεύω πως πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί πάρα πολύ στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή. Και γενικότερα, αρχίζει να γίνεται πραγματικό πρόβλημα και για όλους τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς, αλλά και για τους εμπορικούς μας εταίρους. Εφτά χρόνια χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με, τον Καναδά. Και αν κατάλαβα καλά από ό,τι διάβασα, η συμφωνία με τον Καναδά πρέπει να τεθεί σε ισχύ τέλος αυτού του χρόνου, αρχή του επόμενου. Σιγκαπούρη, εννέα χρόνια έχουν περάσει και ακόμα δεν ξέρουμε πώς να προχωρήσουμε, τι θα γίνει με τις δεσμεύσεις που έχουμε κάνει όσο για τις Ηνωμένε Πολιτείε, το 2014 έγινε 15, 16 και για να είμαστε και ρεαλιστές, μάλλον ούτε τότε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πραγματικά να σκεφτεί όλες αυτές τις λεπτομέρειες και να δει πώς μπορεί να συντομεύσει τη διαδικασία. Έπειτα, ο κύριος ε, Μπαγκουάτη μας προειδοποιούσε για αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει τώρα στην ε, παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η παγκοσμιοποίηση υπάρχει και εκεί και σίγουρα χρειάζεται μεταρρύθμιση των κανόνων ε, για, την, για, την, για τον, χώρο προέλευση, τόπο προέλευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι δεν πρέπει να μείνει μόνο στα λόγια, αλλά να δώσει πράξεις με ουσία. Γι' αυτό χρειάζεται να συζητηθεί ιδιαίτερα μαζί τους για το πώς ακριβώς θα ε, μεταρρυθμιστούν οι κανόνες ε, για την πρόελευση. Έπειτα, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έχουμε διεξάγει πάρα πολλές συζητήσεις για ε, τις επενδύσεις. Τώρα υπάρχει το BIT, αυτό το νέο μοντέλο, αλλά πιστεύω πως χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Διότι εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό νέο ε, μοντέλο για τις επενδυτικές συμφωνίες, πρέπει να ξεφύγουμε από τα παλιά. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με τον Καναδά. Δεν θα αναφερθώ στη Σιγκαπούρη προς το παρόν αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, να δούμε τι συμβαίνει με την Mercosur και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μοντέλα ως βάση για ένα νέο σύστημα, για ένα νέο μέσο. Και αυτό είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέταρτον και τελευταίο, Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στη μεταρρύθμιση των TDI ε, και είναι πράγματι κάτι με το οποίο συμφωνώ. Ωστόσο πιστεύω πως είναι σημαντικό να είμαστε και ρεαλιστές. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις μας με την Κίνα στο άμεσο και προσεχές μέλλον. Θέλουμε μεταρρύθμιση, όμως η πιθανότητα του να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα χαροποιήσει την πλειοψηφία και αυτής της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γενικότερα και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ικανοποιήσει και την Κίνα όσον αφορά την ε, τήρηση του πρωτοκόλλου του ΠΟΕ μέχρι το Δεκέμβριο δεν νομίζω ότι είναι τόσο εφικτό. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς νομίζω πως θα έχουμε προβλήματα με την Κίνα εκεί περίπου στο Δεκέμβριο. Και μάλιστα αν σκεφτούμε και τα προβλήματα με τη Ρωσία, τότε ίσως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ή να επανεξετάσει τη στρατηγική της. και αυτό σε περίπτωση φυσικά που δεν θα καταφέρουμε μέχρι το Δεκέμβριο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλους μας. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω και θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο να ξαναδούμε τη συζήτηση, γιατί άκουσα κάποια ενδιαφέροντα πράγματα εδώ στην Επιτροπή. Να απαντήσω στην κυρία Ντεσαρνέζη, η οποία λέει ότι θα πρέπει να είναι με ένα μέσο η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και όχι σκοπό, αυτός σκοπός. Νομίζω, κυρία Ντεσαρνέζη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση ελευθέρων συναλλαγών βάσει του άρθρου 206 της Συνθήκης που ζητά την άρση των δασμολογικών φραγμών. Εσείς λοιπόν που υποστηρίζετε την Τινησία με τόσο σθένος, ε, να σας πω ότι σήμερα ε, όλα αυτά γίνονται εις βάρος των ε, Ιταλών ελαιοπαραγωγών, για παράδειγμα. Να πω στην κυρία Ρέντινγκ ε, ότι συμφωνώ μαζί της ότι πρέπει να επιβάλλουμε γεωπολιτικούς κανόνες. Πράγματι, νομίζω ότι η συζήτηση είναι λίγο, έχει παρεκτραπεί λίγο. Σήμερα θα πρέπει να δούμε τι έχουν συνεισφέρει τα κράτη-μέλη, κυρίως όσον αφορά την κυριαρχία των κρατών μελών, ακόμα και αν τα κράτη-μέλη χώρισαν την κυριαρχία τους και έδωσαν εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνάψουν συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών, ε, σήμερα τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δείτε για παράδειγμα την περίπτωση της Γεωργίας ιδίως ε, στα θέματα των ε, προστατευόμενων ε, γεωγραφικών ενδείξεων. Από τη μια υπάρχουν οι παραγωγοί, από την άλλη οι χώρες εισαγωγής και φυσικά υπάρχει ανίσως τρόπος ανάπτυξης και ζήτησης μεταξύ των κρατών. Επομένως, κατά την ύποψη μου υπάρχει μια συμβατότητα και αδυναμία να καταλήξουμε σε συνένεση για να έχουμε μια συνολική πολιτική για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Επίσης, να σας πω ότι ε, οι συνέπειε είναι σαφέστατε σήμερα και θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Κανένας δεν τις συζητάει. Σήμερα δυστυχώς αυτές οι συνθήκες ελευθέρων συναλλαγών ε, που θα έπρεπε να είναι καινοτόμε ε, και θέλει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελικά η περιοχή στην οποία υπάρχει η μικρότερη ανάπτυξη σε, από όλες τις περιοχές του κόσμου και μάλιστα η Ευρωζώνη είναι η περιοχή ε, στην οποία υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας. Αν θέλετε να το δείτε, να σας πω απλώς ότι σήμερα αυξάνεται συνεχώς ο λογαριασμός και αρχίζει να χάνει την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου ε, πολίτη. Επομένω, θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα, ακόμα και αν δώσουμε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπραγματευτεί τι συμφωνίε, δεν ξέρουμε κατά πόσον δεν θα, θα πρέπει να συνεχίσει να μην εμπλέκει και τα κράτη-μέλη σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Προύστ. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, Δύο λόγια για να μην επιβαρύνω τη συζήτηση βέβαια, να απαντήσω σε αυτά που μόλις ακούσαμε για το, όλα τα κακά τα οποία θα μας επιφάρει η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και η, η ιδέα ότι είναι κάτι αρνητικό. Υπάρχει μια συμφωνία η οποία συνάφθη πριν από τρει χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με την Νότια Κορέα που κάποτε λέγαμε ότι ε, θα καταστρέψει τις γέφυρες ε, και θα καταστρέψει την αυτοκινητοβιομηχανία μας ε, αυτό που αποδεικνύεται σήμερα είναι ότι αν έχει γίνει κατάλληλη διαπραγμάτευση και έχουμε μια συμφωνία από την οποία βγαίνουν και δυσμένοι όλοι, μετά από τρία χρόνια όχι μόνο έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά έχουμε και ε, πολύ καλό εμπορικό ισοζύγιο. Ε, δύο λόγια μόνον και το έλεγα τότε που είχαμε επίτροπο τον κύριο Εντεχούχου, το οποίος ε, είχε έπασχε από την νόσο αυτή του να τα βλέπει όλα κατά γράμμα ε, πιστεύω ότι οι συμφωνίες πρέπει να γίνονται σεβαστές και επομένως όχι μόνο να προσπαθούμε ε, να συνάπτουμε συμφωνίες οι οποίες να είναι κατάλληλες και επίκαιρες αλλά να υπάρχουν και ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για να μπορούν να ελέγχουν αυτές τις συμφωνίες ώστε να ε, χρησιμοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν όλα αυτά τα μέσα. Για παράδειγμα βλέπουμε τι κάνουν οι ΙΠΑ και πώς αντιδρούν ε, πόσο γρήγορα. Αν υπάρχει κάτι σε δύο μήνες έχουν αντιδράσει. Εμείς θέλουμε εννιά μήνες και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επομένως ε, πρέπει να ε, υπάρχει και η άσκηση του νόμου εξελαχίστων. Υπάρχει μια συμφωνία που έγινε την Παρασκευή και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που είναι κατά, ενώ οι ΙΠΑ θέλουν να βάλουν ε, ε, φορολογία στο 200%, εμείς βάζουμε φορολογία στο 15% που δεν βοηθούν καθόλου και δεν υπάρχει και καμία αξία ε, τιμωρητική. Ουσιαστικά εμείς δίνουμε κίνητρα στους ανθρώπους για να κλέψουν γιατί είναι ελάχιστο αυτό το οποίο θα πληρώσουν, θα πληρώσουν αυτό το οποίο θα πλήρωναν στην πηγή. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να είμαστε εμείς οι αφελείς ως Ευρώπη, ίσα ίσα το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να γίνεστε στη συναισθή Ευρώπη και επίσης κάτι τελευταίο, εδώ θα συμφωνήσω ε, με τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις και ότι είπε ο συνάδελφος. Η γεωργία δεν θα πρέπει να είναι συνεχώς η μεταβλητή προσαρμογής, όπως για παράδειγμα στη Συμφωνία για τη Μερκοσούρη σε άλλες συμφωνίες, γιατί θέλουμε κάθε φορά να έχουμε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και δεν έχουμε καμία εικόνα για το σύνολο και όλα αυτά μπορεί να αποβούν εις βάρος της γεωργίας μας και Εάν δεν δούμε ότι το σύνολο είναι απλώς μια προσαρμογή στη δυνατότητα ε, να έχουν και ε, επικερδείς ε, τομείς και στη γεωργία, θα χαθεί η γεωργία και η παραγωγή μας. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φόλμπραχ τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώ ε, συζητάτε αυτή τη στιγμή τι τροπολογίε που έχετε υποβάλει για την έκθεση τη κυρία Μπεγκίν. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κάνω και εγώ κάποιε σύντομε παρατηρήσει. Πρώτον, όσον αφορά τι παρατηρήσει του κυρίου Κάσπαρη. Είναι πολύ θετικό να λέμε πάντα ότι το εμπόριο είναι πολύ θετικό για την οικονομική ανάπτυξη και για του ίδιου του καταναλωτέ. Αυτό άλλωστε το έχουμε και στα πλαίσια τη πρωτοβουλία Εμπόριο για Όλου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή την άγουσα ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τα όσο είπε κύριο Μάρτιν για τον, το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας, σαφώς το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα πολιτικό και εξετάστηκε και σε στο πολιτικό επίπεδο τις τελευταίες αυτές μέρες. Επομένως εκεί πέρα θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση, το υψηλό δηλαδή πολιτικό επίπεδο. Είπατε επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμόζονται οι συμφωνίες αυτές και αναφερθώ και στα είπε ο κύριο Στάκουλα για τους πόρους και για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Αυτή τη στιγμή όντως υπάρχουν πάρα πολλές εμπορικές συμφωνίες οι οποίες εκκρεμούν και επομένω όντω χρειαζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερου εργαζομένου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι συμφωνίε αυτέ. Όσον αφορά το ζήτημα τη αναθεώρηση, θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πλέον ένα σύστημα ετήσιο για την αναθεώρηση και αξιολόγηση των εμπορικών συμφωνιών που θα αρχίσει να λειτουργεί από του χρόνου και κατά αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε και τις συμφωνίες αυτές οι οποίες θα πρέπει να εξολογηθούν και κατά το δεύτερο ήμιση του 2017. Κάποιες άλλες σύντομε παρατηρήσεις. Η κυρία Μακλάρκιν ανεφέρθηκε στη βιοπικιλότητα, το σημειώνουμε αυτό. Η κυρία Ρέντιγκ και ο κύριος Στάκουλ επίσης ανέφεραν τη σημασία της ψηφιακής οικονομίας μεταξύ άλλων. Πρέπει να σας πω ότι το θεματολόγιο για την περίοδο μετά του Ναϊρόμπι ασχολείται ιδιαίτερα με τα ψηφιακά ζητήματα. Τα συζητάμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο, ο κυρία Αργεντίνη και ο κύριο Σόλτ αναφέρθηκαν σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δοντολογικό εμπόριο, το δίκαιο εμπόριο και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων. Συμφωνούμε με τι παρατηρήσει σα και χαιρόμαστε που έχετε υποβάλει τέτοιε τροπολογίε. Στα πλαίσια τη στρατηγική εμπόριο για όλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να φωτίσουμε και αυτέ τι διαφορετικέ διαστάσει και όχι μόνο τι πιο παραδοσιακέ διαστάσει που έχουμε στα πλαίσια τη εμπορική πολιτική. Να δώσουμε τέλο το λόγο και στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους ε, για αυτή την πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Σίγουρα πολλά από τα πράγματα τα οποία είπατε έχουν ληφθεί υπόψη. Να ευχαριστήσω επίσης και τους κοιόδες ε, για με τους οποίους έχουμε ένα πολύ θετικό διάλογο. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ μπορούσα να ακούσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους συνεδρίαση αυτή και απευθύνομαι κυρίως αυτούς διότι αυτοί δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών και είναι σημαντικό λοιπόν να ακούγονται και οι δικές τους απόψεις. Έχουμε ήδη λάβει υπόψη μας πολλές από τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σήμερα. Αναφέρομαι στην κυρία Ρέντινγκ για παράδειγμα, με την οποία συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία είπε στη δική της την παρέμβαση. Αναφέρουμε για παράδειγμα το ζήτημα της εντολής, την συμβαστική τροπολογία 13. Οι τελευταίες αυτές συμβαστικές τροπολογίες διανεμήθηκαν δυστυχώς μόνο σήμερα το πρωί, επομένως ενδεχομένως δεν είχατε τον χρόνο να τις διαβάσετε. Και αναφέρομαι επίσης και στη συνάδελφο Ροντρίγκε με τη βοήθεια τη οποία έχουμε καταφέρει να εντάξουμε πολλέ από τι παρατηρήσει τη στι συμβαστικέ τροπολογίε, ιδίω τα όσα είπε για τη διάσταση του φύλου, ζήτημα με το οποίο ασχολείται και ο συνάδελφο Σόλτ. Επεξεργόμαστε το ζήτημα αυτό και θα συμπεριληφθεί κατά πάση πιθανότητα στην τροπολογία 12. Όσον αφορά επίση τη συμβαστική τροπολογία 21, εκεί θα γίνεται μία αναφορά και στη δική σα τροπολογία που αφορά τι χώρε του Μερκοσούρα με την κυρία Ντεσσαρνέτς. Συμφωνώ μαζί της ότι όντως το εμπόριο θα πρέπει να αποτελεί απλώ ένα μέσο και σε καμία περίπτωση έναν αυτοσκοπό. Αυτό άλλωστε το λέω και στην αρχή της έκθεσής μου. Στο σχέδιο έκθεσής μου αναφέρω στο προήμιο ακριβώς το ζήτημα αυτό. Και όσον αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα, θα φροντίσουμε όντω να αφήσουμε εκτό τον τομέα αυτό από τι εμπορικέ συμφωνίε. Εν γέννη, μπορώ να πω ότι θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε όλε αυτέ τι ιδέες που ακούσαμε αυτή τη στιγμή από τους συναδέλφους. Συμφωνώ επίσης ε, με τον κύριο Ντάνιελ Κάσπαρη στα όσα είπε, δηλαδή ότι θα πρέπει η έκθεση αυτή να γίνει όσο δυνατόν πιο απλή, πιο συνοπτική και ότι θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στα πιο σημαντικά ζητήματα προκειμένου να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τις θέσεις που θέλει να προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι έχουμε να καλύψουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας και βρισκόμαστε, θεωρώ, στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία λοιπόν θα γίνει τον Ιούνιο, θα γνωμοδοτήσουν και άλλες επιτροπές. και πιστεύω πως θα έχετε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να διαπραγματευτείτε τις συμβαστικές τροπολογίες. Επόμενα σημεία, 7 και 8, είναι μια κοινή συζήτηση για την κατάσταση στο Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία. και για τις κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν. Η κυρία Τσάκη, συγγήτρια, δυστυχώς δεν βρίσκεται εδώ. Αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Τάκουλα για να μας ενημερώσει εκ μέρους της. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά πρόεδρε, θα μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Χάκε, η οποία δυστυχώς λείπει σήμερα. Η γνωμοδότηση αυτή στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αφορά τις ε, πτυχές της ευρωπαϊκής ε, στρατηγικής για το Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία η οποία επεγράφει πέρυσι. Μέρος της πυρηνικής συμφωνίας με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεχτήκαμε να άρουμε όλες τις εκκυρώσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί δυνατότητα να ανοίξουν εκ νέου οι αγορές του Ιράν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μετά από πολλά χρόνια αυτοαπομόνωσης, η οικονομία του Ιράν έχει ανάγκη επενδύσεις. Έχει ανάγκη επενδύσεις και ο πληθυσμός του Ιράν που είναι ε, σχετικά υψηλά, ε, σχετικά μορφωμένος, μπορεί να υποφεληθεί από αυτό. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις αυτές θα συνοδευτούν και από ουσιαστικές βελτιώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει τη θέση της έτσι ώστε να πιέσει για να εφαρμοστούν αυτές οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών του Ιράν να βελτιωθούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των γυναικών και το δικαίωμα ελεύθερων και ανεμπόδιστων εκλογών. Είναι μερικά παραδείγματα μόνο. Επιπλέον, τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να υπάρξει ένας πραγματικά ιδιωτικός τομέας. Έχουν γίνει σίγουρα ε, πολλά τα οποία καθιστούν πιο δύσκολη την σύναψη πορικών σχέσεων με το Ιράν. Όμως ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις πιθανότητες επανεκκίνησης των ε, συνομιλιών ε, σχετικά με την προσχώρηση του Ιράν στον ΠΟΕ, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα ενσωματώσει τη χώρα στο παγκόσμιο σύστημα και θα την κρατήσει υπόλογη για τις πράξεις της και θα την καλέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Αυτά λοιπόν από εκ μέρους της εισηγήτριας και θα χαρώ να ακούσω τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Προύστ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή τη γνωμοδότηση, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ ισορροπημένη και αναφέρεται και σε θέματα τα οποία μέχρι πρότινος ε, τα υποτιμούσαμε, ε, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, η ανάγκη για τις υποδομές, ε, η απελευθέρωση του ορίου ηλικίας, γιατί αυτά μας δίνουν δυνατότητες σε εμπορικό επίπεδο. Εδώ στη γνωμοδότηση αναφερόμαστε μεν στις εμπορικές σχέσεις, αλλά νομίζω ότι η συντάκτρια ανέφερε με πολύ ευφύ τρόπο το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο και που εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέμε όλοι και νομίζω ότι πρέπει ε, να το πούμε γιατί το Ιράν ε, έχει εξαιρετικές δυνατότητες μεν για τις επιχειρήσεις μας, αλλά και γιατί πρέπει να θεμελιώσουμε εκ νέου και σχέσεις οι οποίες πηγαίνουν πέραν του εμπορίου και αφορούν τον πολιτισμό μας, ε, τις ανταλλαγές, αλλά και τη διπλωματία τούτου δεδομένου, προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτές τις χώρες, πρέπει οι επιχειρήσεις μας ε, να ε, μπορούν να νιώθουν εμπιστοσύνη. Αναφερόμαστε και στην προφορική ερώτηση που έχουμε, διότι αναφερόμαστε σε πάρα πολλές αβεβαιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας, λόγω ε, το, της διαφθοράς, ε, τη ρευστότητα και τα ε, αδυναμίες πληρωμών. Νομίζω ότι οι σχέσεις μας θα πρέπει να είναι σχέσεις εμπιστοσύνης. Ε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις εμπορικές σχέσεις της περιοχής. Εγώ ήμουνα μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο στο Κατάρ για να συζητήσω ε, τα θέματα της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες. Αλλά ε, αλήθεια είναι ότι η επανέναρξη των εμπορικών σχέσεων με το Ιράν θα αλλάξει τις γεωπολιτικές σχέσεις, κυρίως με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ε, που μπορεί να έχουν προβλήματα λόγω των συναλλαγών ε, και των πληρωμών και θα μπορούσαν ίσον μεν να παίξουν το ρόλο του τραπεζίτη, αλλά αν λάβουν να παίξουν το ρόλο του, του τραπεζίτη θα έχουν και ε, κυρίαρχη άποψη για την επιλογή του πελάτη. Επομένως θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ποιότητα της γνωμοδότησης, τη συντάκτρια και φυσικά το ΕΛΚ θα επιδείξει επικοδομητικό πνεύμα σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τη συντάκτρια της γνωμοδότησης για τα πολύ θετικά στοιχεία που έχει το σχέδιο γνωμοδότησής της. Η συμφωνία που συνάφθηκε πέρσι με το Ιράν για τα πυρηνικά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Όλοι θα υποφεληθούν αν το Ιράν είναι υπεύθυνο μέλος της διεθνούς κοινότητας και θα διευκολύνουν την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή εάν δράσει βάσει και της συμφωνίας που υπέγραψε και δείξει και καλή διάθεση για την εφαρμογή του περιεχομένου συμφωνίας. Είναι πολύ ψηλά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Ιράν. Ας δούμε άλλωστε και τις αντιπροσωπείς υψηλού επίπεδου που επισκέφθηκαν την Τεχεράνη τους προηγούμενους μήνες. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σίγουρα μπορούν να επωφεληθούν. εάν εφαρμοστεί καταλήλως το στρατηγικό έγγραφο για τις σχέσεις με το Ιράν. Αλλά εδώ να κάνω έκκληση, γιατί πρέπει να συντονίσουμε την πολιτική μας για το Ιράν, με την εξωτερική πολιτική, τα θέματα ασφαλείας και τις δεσμεύσεις του εξωτερικού εμπορίου. Δεν μπορεί να είναι μια κοντόφθαλμη προσέγγιση γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος να χάσουμε τον όλο στόχο των σχέσεων με το Ιράν. Σίγουρα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις του ε, για μια αμφίδρομη διαδικασία και μάλιστα το αναφέρει και η συντάκτη της γνωμοδότησης ρητός. Ε, υπάρχει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητούνται κάθε φορά με το Ιράν. Η δεύτερη σημαντική διάσταση, την οποία ανέφερα, αναφερόμαστε στην περιφερειακή διάσταση και το πόσο περίπλοκες είναι οι σχέσεις μας με το Ιράν. Αυτό μπορεί και πρέπει να είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά είναι, αν είναι πολύ μεγάλη διμερής διάσταση στις σχέσεις μας με το Ιράν, ελοχεύει ο κίνδυνος να επιδενώσουμε τις σχέσεις μας με άλλους περιφερειακούς παράγοντες, είτε από το μουσουλμανικό κόσμο, είτε από τον υπολείπους. Πρέπει να ε, προσέξουμε ιδιαίτερα την πολύ περίπλοκη παραπραγματικότητα που επικροτεί στην περιοχή για να έχουμε και τα ωφέλη που περιμένουμε. Το Ιράν λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσει τις ε, πολιτικές αυτές και τη συμφωνία και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα, αλλά να συνεισφέρουμε και στη βελτίωση της ευημερία και τη καλή διακυβέρνηση στο Ιράν. Όχι μόνο οι επιχειρήσεις και το χρήμα, αλλά και τις ε, σχέσεις με το Ιράν, αλλά πρέπει να δούμε και τις ε, συμμετρικά εποφελείς διαδικασίες. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα με το Ιράν, διότι θα δώσει μία όθηση στην ε, ε, πιεσμένη οικονομία του Ιράν και θα επιτρέψουμε να επανενωθεί με τον κόσμο εν γέννη το Ιράν και να υποφεληθεί ε, από τους τεράστιους ε, φυσικούς πόρους που έχει, ξεκινώντας από την ενέργεια. Εδώ βέβαια πρέπει να προσέξουμε και τη διαφθορά και την ανάγκη να εφαρμόσουμε ένα αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα, να υπάρχει μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα και να ε, υπάρξει προστασία του επενδυτικού κεφαλαίου, ιδίως σε σχέση με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βεβαίως και μεγαλύτερη διαφάνεια. Κατά την άποψή μου, εκεί που θα πρέπει να προσδώσουμε σημασία είναι να συζητήσουμε ε, σαφώς τα θέματα ενέργειας με το Ιράν, γνωρίζοντας ότι υπάρχει και η Ενεργειακή Ένωση, που είναι μία από τις ουσιαστικές πτυχές που μας αφορούν. Θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση από έναν και μόνο πάροχο και θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικέ πηγές και οδούς ε, παροχής ενέργειας. Το Ιράν μπορεί να είναι ένας από τους δυνητικούς εταίρους μας και για να υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και να μπορέσουμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του Ιράν θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί της η Ευρώπη ώστε να μπορέσουμε να ε, βοηθήσουμε και την προσχώρηση του Ιράν στον ΠΟΕ. Όσον αφορά τις κυρώσεις και εδώ ε, νομίζω ότι η πολιτική μου ομάδα ε, συμμετέχει στις κοινέ προσπάθειες. Ε, θα πρέπει να συζητήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι κυρώσεις που απομένουν για το Ιράν δεν θα αποτελέσει επιπλέον πρόσκευμα για τις επιχειρήσεις μας. Ε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και επομένως η ομάδα μου θα υποστηρίξει άνω φόρων την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία για να έχουμε μια ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση στην έκθεσή μας για το Ιράν. Για το ECRM, Ευχαριστώ. Εγώ αντικαθιστώ τον David Campbell, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για την έκθεση αυτή. Η ομάδα του ECR μπορεί να συμφωνήσει με τα περισσότερα σημεία του σχεδίου αυτού γνωμοδότησης προς την ΑΦΕΠ όσον αφορά τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράν σε συνέχεια τη Πυρηνική Συμφωνία, ιδίω όσον αφορά τι νέε ευκαιρίε που δίνονται για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, επιχειρήσεις με συγχωρείτε, και για την μείωση αυτή της οικονομικής απομόνωσης του Ιράν, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί να ωφελήσει και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούμε πάντω ότι ενδεχομένω να μην πρέπει αυτή τη στιγμή να αρθούν άλλες κυρώσει που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τη δημοκρατία ή με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έχουμε ως προς αυτό κάποιο πρόβλημα διαβάζοντας το σχέδιο της γνωμοδότησης και διαβάζοντας και το προφορικό σας ερώτημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδίως ενώψη οποιασδήποτε ψηφοφορίας. Ο κύριος Μπούκνερ. Ευχαριστώ πολύ. Δίχως αμφιβολία αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Ιράν είναι ότι η ε, πολίτες του Ιράν επιζητούν μια αλλαγή. Μια αλλαγή από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι το πιο αποτελεσματικό μέσο ε, αντιμετώπισης είναι όχι η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Ιράν, όχι δηλαδή να δείχνουμε με το δάχτυλο τη διαφθορά και τα λάθη τα οποία ε, παρατηρούμε, αλλά η προσπάθεια να συζητήσουμε στο ίδιο επίπεδο με την κυβέρνηση του Ιράν. Γι' αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Σχάκη για αυτό το πάρα πολύ καλό σχέδιο έκθεσης. Πιστεύω πως πολλές επιτυχίες από αυτό το σχέδιο είναι ε, και θα έπρεπε να τις... Ε, στηρίξουμε. Εμείς ως Ευρωπαίοι δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε τους ηθικολόγους, διότι έχουμε πολλά δικά μας προβλήματα και θα έπρεπε ιδιαίτερα στον τομέα της διαφθοράς να αναλογιστούμε τι ε, έχουμε κάνει. Βλέπε Panama Papers. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να δείχνουμε το δάχτυλο όταν έχουμε τη δικιά μας βολιά λερωμένη. Πιστεύω λοιπόν πως οι κυρώσεις και η άρση των κυρώσεων δεν θα επιφέρουν κάποια βελτίωση στην κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η άρση των κυρώσεων ως αποτέλεσμα της πυρηνικής συμφωνίας δεν έχει προϋποθέσεις. Όμως, αφήνοντας αυτές τις κυρώσεις, εάν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι, πιστεύω πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ίση αντιμετώπιση προς την κυβέρνηση του Ιράν. Έτσι μόνο θα καταφέρουμε να ασκήσουμε πίεση για να βελτιωθεί η κατάσταση για τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπορέλη, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο τις διπλωματικές νέες αυτές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν, τις οποίες θα πρέπει να χαιρετήσουμε, καθότι συμβάλλουν στην καλύτερη ισορροπία, όχι μόνο πολιτική, αλλά και εμπορική της όλης περιφέρειας αυτής. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό η δική μας η Επιτροπή να ασχοληθεί με το γενικότερο αυτό πλαίσιο το οποίο η κυρία Μογκερίνη ονόμασε διπλωματία, η οποία δεν θα έχει να κάνει μόνο με την πολιτική, αλλά θα έχει να κάνει επίσης και με τη συνεργασία. Και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπληρώνεται η στρατηγική αυτή με περισσότερα στοιχεία συνεργασίας. Είναι σημαντικό λοιπόν η προσέγγισή μας να είναι σφαιρική απέναντι στο Ιράν και να μην περιοριστεί σε συγκεκριμένου μόνο εμπορικού τομεί. Πέρα από την οικονομική διάσταση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να στηρίξει και κάποιες θεμελιώδεις αξίες και να προωθήσει κάποιες θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες στις σχέσεις που έχει με το Ιράν. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πραγματικά ένα στρατηγικό πλαίσιο όσον αφορά την εμπορική μας σχέση με το Ιράν. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να έχουμε ισχυρές βάσεις με ένα συγκεκριμένο μελλοντικό προσανατολισμό. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε ξεκάθαρα και προ τι Ηνωμένε Πολιτείε και ρωτώ ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσονται και διαπραγματεύσει για το TTIP ότι ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι σαφώ ο σημαντικότερος μας εταίρος, αλλά είναι πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να έχουμε μια κάποια εμπορική και οικονομική αυτονομία. Θα ήθελα να ελπίζω ότι μπορούμε να εμβαθύνουμε και στα σημεία αυτά κατά την επεξεργασία του σχεδίου γνωμοδότησης. Um, um, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους συνδέλφους για τα σχόλιά τους, με τα οποία σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Μου κάνει εντύπωση η τελευταία έκθεση της Amnesty International όσον αφορά την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια του Ιράν. Η γνωμοδότηση και το προφορικό ερώτημα προφανώς είναι αρκετά ισορροπημένα, αλλά τίθεται και ένα γενικότερο θέμα. Πώς η εξωτερική μας δράση και η εμπορική μας δράση χρησιμοποιείται τελικά για να προωθήσει ή όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες εταίρους ή δυνάμει χώρες εταίρους. Και εδώ επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο Ιράν. Ας μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι η μόνη χώρα όπου εκτελούνται περισσό, που έχουν εκτελεστεί οι περισσότεροι άνθρωποι πέρυσι και έχουμε και την Κίνα βέβαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν σαφώς προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε επικεφαλής ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων που δέχονται απειλές ή φυλακίζονται. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και του συνέχερστε, το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και γενικότερα έχουμε μια κατάφορη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει στο κείμενο της γνωμοδότησης, κάθε φορά που λέμε για μία ενδεχόμενη ανανέωση των εμπορικών μας σχέσεων με το Ιράν, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ανησυχία που έχω είναι ότι στις πρόσφατε υψηλόβαθμε αντιπροσωπείε που πήγανε στο Ιράν, η πληροφορία που μα ήρθε είναι ότι σε ορισμένε περιπτώσει παραμερίζονται τελικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπερτερούν, επικρατούν άλλα συμφέροντα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε διαφορετικά τη σχέση μα με του εταίρου και ιδίω με αυτό τον εταίρο, με το Ιράν. Θα ήθελα να το το ζήτημα αυτό. Συμφωνώ με αυτά που είπαν και οι εκπρόσωποι και ο εκπρόσωπο πολιτική μου ομάδα. Θεωρούσα πάντω θα πρέπει να τονίσω κάπω περισσότερο. Κυρία Ντεσαρνέζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρεται εδώ. Αλλά θα πρέπει από αυτή την άποψη ε, αυτή στιγμή βάλουμε και το Ιράν στο παιχνίδι να μπορέσουν οι προοδευτικοί να κερδίσουν το θέμα αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εξού και οι αμερικανικές κυρώσεις. Αν εμποδίζουν οποιαδήποτε οικονομική ανάπτυξη, οποιαδήποτε επένδυση στο Ιράν, αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν το άνοιγμα θα είναι οι προοδευτικοί ένα, αλλά θα υπαναχωρήσουν ε, προς όφελος των πιο ακραίων και συντηρητικών στοιχείων. Επομένως, σας ευχηστώ την προσοχή είναι πάρα πολύ προβληματικό το θέμα αυτό των Αμερικανικών κυρώσεων, εάν τελικά δεν επιτρέψουν στους Ιρανούς να υποφεληθούν από τις αλλαγές και μάλιστα ε, τις πολύ συγκεκριμένε αλλαγές ε, από την άρση του εμπάργου. Αλλιώς σε επόμενους ε, μήνες θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε ότι αυτή ήταν η καλή πολιτική απόφαση. Είναι πολύ προβληματικό το θέμα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική προφορική ερώτηση ακριβώς για αυτό το λόγο. Ε, σίγουρα το Ιράν θα πρέπει να ξαναμπεί στο παιχνίδι ε, και ε, είναι προς το συμφέρον μας οι προοδευτικοί να κερδίσουν έδαφος στο Ιράν. Χρειαζόμαστε το Ιράν, να μην το φτυλισμονούμε, για να μπορέσουμε να έχουμε και μια κατάλληλη πολιτική για τα όσα συμβαίνουν στη Σύρια. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ και εγώ στις συμφωνίες της Γενέβης, ε, τις υποστηρίζω και εγώ γιατί επιτρέπουν ε, στο Ιράν ε, να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο κύριος Φεράν. Αλλά βέβαια εδώ υπάρχει το θέμα των αμερικανικών ε, δικαιωμάτων και επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε αρνούνται να εκφράσουν την άποψή τους για αυτό το οποίο απαγορεύουν, οι τράπεζες έχουν παραλύσει σε θέματα επενδύσεων προς το Ιράν, διότι οι αμερικανικές κυρώσεις θεωρητικά αφορούν ακόμα τον, την τρομοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και υπάρχει ένας εταίρος ο οποίος πλήττεται από το θέμα αυτό, η Airbus, διότι δεν έχει τράπεζες να την υποστηρίξουν. Βλέπω επίσης ότι υπάρχει πρόοδος ε, με το Ιράν, αλλά ο μεγάλος απόν από τη συζήτηση είναι η Ρωσία. η οποία πιστεύω ότι θα μπορούσε να συμμετέχει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για έναν εταίρο ο οποίος θα λείψει πάρα πολύ από την Ευρώπη. Ο κύριος Προύστ. Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα καταλάβει ότι μπορούμε να παρέμβουμε τώρα και για την προφορική ερώτηση. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω από αυτά που είπε η κυρία Ντεσαρνές, γιατί νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υποστήριξε το ΕΛΚ αυτή την ε, ε, προφορική ερώτηση. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Όπως και σε άλλες περιοχές βλέπουμε τη συμπεριφορά των Αμερικανών. Ε, έχουν λόγους πάντα να παρεμβαίνουν, είτε θέματα ασφαλείας, είτε γεωπολιτικούς ε, ε, και θέτουν θρένο στις επενδύσεις και στις ανταλλαγές. Αλλά το πρόβλημα τελικά είναι ότι τους αφορά και τους ίδιους. Και βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μας έχουν εξαιρετικές δυνατότητες, αλλά το είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, υπάρχει θέμα εμπιστοσύνη τρία προβλήματα ε, κατά την άποψή μου ε, ε Τα είπατε και εσείς και η κυρία και άλλοι. Το ε, θέμα το εδαφικό του Αμερικανικού δικαίου. Και υπάρχει και το θέμα του να μην μπορεί να γίνουν σήμερα συναλλαγές σε ευρώ. Υπάρχει περίπτωση της BNP Paribas στη Γαλλία που τη γνωρίζουν όλοι, η τράπεζα τελικά τιμωρήθηκε γιατί έκανε συναλλαγές σε δολάρια και το πρόστιμο είπατε ήταν υπερβολικό και ανερχόταν σε 9 δις ευρώ, ε, δολάρια, συγγνώμη και αυτή τη στιγμή οι επενδυτές είναι τρομοκρατημένοι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν μπορούμε να θέσουμε το ευρώ στο επίκεντρο των ε, διαπραγματεύσεων για εμπορικά θέματα. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, τρίτον, πρέπει να έχουμε την ίδια ανάλυση με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή που ήρθε, ήρθε το εμπάργκο για τις κυρώσεις για τα πυρηνικά θέματα, ε, υπάρχουν ε, όμως ε, το πρόγραμμα για τους βαλιστικούς πυράβλους, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα με το Ιράν. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζουμε και τίθεται και το ερώτημα σήμερα αν μπορούμε να επενδύσουμε στο Ιράν. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις επενδύουν και νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία σε αυτό και υπάρχουν οι κυρώσεις κατά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που είναι διάκριση. Θεωρώ λοιπόν ότι η περίπτωση αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκη ε, αδελφοκτονία με τις Ηνωμένε Πολιτείε και νομίζω ότι όπως και οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες, το ΑΕΛΚ θα περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε και τι συνέχεια θα δώσουμε στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φίνη από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Ρέι. Είμαι μαζί με τον κύριο Φραντσέσκο Φίν. Είμαστε και οι δύο από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και θα απαντήσουμε και οι δύο ε, στις ερωτήσεις για τις κυρώσει. Εγώ θα ολοκληρώσω με σχόλια για την γενικότερη στρατηγική για το Ιράν. Καταρχά σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου μας δώσατε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για μια έκθεση σχετικά με τη στρατηγική για το Ιράν και αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Θα ήθελα, εν συντομία, να σας αναφέρω τη στρατηγική μας, τη μελλοντική μας στρατηγική για το Ιράν. Στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Καταρχάς, την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της πυρηνικής συμφωνίας, μια συμφωνία η οποία ήταν η βάση ακριβώς την οποία χρησιμοποίησαμε για ε, να ανοίξουν οι διαβουλεύσεις με το Ιράν. Η εφαρμογή της λοιπόν πλήρως είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η διαδικασία. Όπως γνωρίζετε, οι Ηνωμένε Πολιτείε παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και έπαιζαν σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και στην διαδικασία εφαρμογής. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, το είπατε εκπρόσωπος, επιβλέπει τις διάφορες ομάδες που ασχολούνται με την εφαρμογή της συμφωνίας. Η εφαρμογή λοιπόν της πυρηνικής συμφωνίας είναι μια πολύ σημαντική διάσταση ε, της στρατηγικής μας έπειτα ανανέωση των διμερών σχέσεων. Και αυτό καθίσταται δυνατό ακριβώς γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας ε, αποφάνθη ότι το Ιράν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Αυτή η διμερής διαβούλευση άρχισε στις 16 Απριλίου, όπου μετέβησαν πολλοί επίτροποι στο Ιράν και η ύπατη εκπρόσωπος ονόμασε αυτό το νέο στάδιο ε, ένα νέο στάδιο διαλόγου, ολοκληρωμένος διάλογος για συνεργασία όπου υπάρχει αμοιβαίο ε, συμφέρον, σημαντικός, αμφιλεγόμενος σε πολλά δύσκολα σημεία, όμως πάρα πάρα πολύ σημαντικός και απαραίτητος. Το όραμα είναι να αρχίσει διάλογος κατά τομής. Καταρχάς συμφωνήσαμε κάθε χρόνο να γίνονται πολιτικές ε, διαβουλεύσεις, να συσταθεί, να δημιουργηθεί μάλλον ένας ε, διάλογος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. και τονίσαμε τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υψηλή θέση που πρέπει να έχουν στις προτεραιότητές μας. Έπειτα, διάλογο σχετικά με τη μετανάστευση, την ενέργεια, την οικονομία και, αυτό αφορά και εσάς, να ενισχύσουμε τους εμπορικούς και επενδυτικούς μας δεσμούς. Και αυτό θα αρχίσει με την στήριξή μας στην προσχώρηση του Ιράν στον ΠΟΕ. Αυτό συμπεριλαμβάνεται και στην έκθεση που ε, συζητάμε. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό το Ιράν να συμμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες και οι ευκαιρίες που προκύπτουν είναι τεράστιες. Μιλάμε για την μεγαλύτερη οικονομία ε, στην περιοχή. Το Ιράν έχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και ε, πετρελαίου. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα εμπόδια που σας ανέφερα, υπάρχει διαφθορά, υπάρχει ε, συγκεντρωτική οικονομία, έλλειψη διαφάνειας, αδυναμίες στον τραπεζικό τομέα και φυσικά αυτά πρέπει να εξεταστούν και να συζητηθούν. Αλλά ο επόμενος πυλώνας είναι αυτό που αναφέρατε πολύ και από εσά. Είναι η συζήτηση με το Ιράν έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί ειρηνική λύση για τις συγκρούσεις στην ε, περιοχή. Καταρχάς, στο θέμα της Συρίας σίγουρα δεν συμφωνούμε με ό,τι κάνει το Ιράν. Όμως χρειάζεται συζήτηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για επίλυση των συγκρούσεων που μαστίζουν την περιοχή. Αυτά λοιπόν εν ολίγη σχετικά με την στρατηγική μας για το Ιράν. Προσπαθούμε δηλαδή να αντισταθμίσουμε τα θετικά με τα αρνητικά έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τώρα τον ε, εξοεδαφικό χαρακτήρα των κυρώσεων των ΗΠΑ, θα αναφερθώ εδώ πέρα στα τρία ερωτήματα τα οποία τέθησαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και εμεί ω υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχουμε αναλύσει και το αναλύσαμε και κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσαμε εκτενέστατα να συζητήσουμε το ζήτημα των εξωεδαφικών επιπτώσεων που έχουν οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τη δική σας την ανάλυση, γιατί οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι εξωεδαφικές εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός του Αμερικανικού συστήματος. Εξαιτίας όμως του ρόλου που δραματίζει το Αμερικανικό οικονομικό σύστημα και οι Αμερικανικές επιχειρήσεις προκύπτει αυτός ο εξεδαφικός χαρακτήρας. Υπάρχει αυτή η εξεδαφική επίπτωση χωρίς αυτή να υφίσταται αυτή καθεαυτή από την αρχή οι εκκρεμούσει αυτή τη στιγμή αμερικανικέ κυρώσει, οι οποίε δεν συνδέονται με την πυρηνική συμφωνία, στα πλαίσια τη οποία είχαμε άλλε κυρώσει, οι κυρώσει των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν λοιπόν με την τρομοκρατία ή με άλλα ζητήματα όπω τα ανθρώπινα δικαιώματα, ουδέποτε αποτελούσαν τμήμα των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων. Και για αυτό το λόγο, μετά το γενικό αυτό κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης δεν ήρθησαν, γιατί θεωρείται ότι ασχολούνται με άλλους τομείς. Άρα, οι Ηνωμένε Πολιτείε μέχρι στιγμής έχουν εφαρμόσει πλήρως τις δικές τους τις δεσμεύσεις όσον αφορά το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, διότι απέσυραν τελικά όλες τις κυρώσεις που είχαν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν όλες τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κυρώσεις που είχαν να κάνουν με το πρόγραμμα αυτό οι εκκρεμούσεις αυτή τη στιγμή κυρώσεις, αυτές που απομένουν, δημιουργούν όντως ένα πρόβλημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της εμβέλειας που έχει το δολάριο και η αμερικανική οικονομία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε δημιουργήσει μια, ένα πολύ συστηματικό σύστημα συνεργασίας με την αμερικανική πλευρά, προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια Προ τι ευρωπαϊκές επιχειρήσει επιχειρήσεις, με συγχωρείτε, ως προ επιπτώσει που έχουν οι αμερικανικές αυτές κυρώσεις. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ήδη δημοσιεύσει κατευθυντήρε γραμμέ όσον αφορά τι κυρώσεις αυτές. Έχουμε συζητήσει με τους Αμερικανούς αυτές τι κατευθυντήρες γραμμές πολλές φορές στο παρελθόν και Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάει στην Ουάσιγκτον και συζητήσαμε αυτές τις ε, κατευθύνες γραμμές προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια, μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το πώς επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Κάνουμε επίσης δύο συγκεκριμένες αποστολές σε σχέση με το ζήτημα αυτό και βασιστήκαμε σε πληροφορίες που μας δίνανε διάφορες αμερικανικές επιχειρήσεις. Αυτές λοιπόν οι κατευθυντήρες γραμμές τροποποιήθηκαν ήδη μια πρώτη φορά, θα τροποποιηθούν και μια δεύτερη φορά μετά τις διαβουλεύσεις που είχαμε με την Αμερικανική πλευρά. Απαντώντας λοιπόν στο ερώτημά σας πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε στενή επαφή με την Αμερική προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη σαφήνεια και διαφάνεια ως προς το πώς επηρεάζονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις. Επίσης ε, γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως ο τραπεζικός τομέας. Παράλληλα όμως μας ενθαρρύνει η θετική εξέλιξη που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να επικρατεί. Προφανώς οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες δεν έχουν καταφέρει να επιστρέψουν και να επενδύσουν στο Ιράν Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν ε, μικρές και μεσαίες τράπεζες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν αυτή τη στιγμή να συνδέονται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά με τράπεζες ε, αντίστοιχου μεγέθους στο Ιράν. Τα πράγματα λοιπόν βελτιώνονται, δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή πρόοδο όσον αφορά τις μεγάλες και με, τις μεγαλύτερες μάλλον ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ήδη κάποιες θετικές επιπτώσεις για τις μικρομεσαίες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότερες τράπεζες του Ιράν επίσης έχουν ενταχθεί στο σύστημα SWIFT. Υφίσταται λοιπόν πλέον το γενικότερο αυτό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να αποκαταστήσουμε τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν. Πρέπει απλώς να περιμένουμε λίγο περισσότερο, αλλά θα πρέπει και το ίδιο το Ιράν να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα σε εσωτερικό επίπεδο προκειμένου να αποκατασταθεί το απαραίτητο επίπεδο εμπιστοσύνη. Το νομικό πλαίσιο πλέον υφίσταται. Η τεχνική πλευρά υφίσταται επίση, για παράδειγμα το σύστημα SWIFT. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη. Και βέβαια αυτό είναι αμφίδρομο. Θα πρέπει να αποκατασταθεί και από την πλευρά του Ιράν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχουν σαφεί επιχειρηματικέ δομέ, έτσι ώστε κάθε φορά που μια ευρωπαϊκή επιχείρηση επενδύει στο Ιράν να μην φοβάται ότι τα πράγματα μπορεί να μην κινηθούν με απόλυτη διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχουν μέτρα κατά της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Πρέπει αυτή τη στιγμή με τα απαραίτητα μέτρα τα οποία θα λάβει το Ιράν να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να δώσουμε απόλυτη αφήνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να πτύξουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο Ιράν, αλλά θα πρέπει αμοιβαία, αμφίδρομα και το Ιράν να δράσει κατά τέτοιο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι αν η άρση των κυρώσεων δεν αποφελήσει τελικά το Ιράν, τότε όλη αυτή η πυρηνική συμφωνία θα τεθεί ένα αμφιβόλο. Ο κύριος Στάκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης ηγητές και όλα τα μέλη της Επιτροπής για τα σχόλιά τους. Θα τα μεταφέρω στον εισηγητή, στην εισηγήτρια. Επίσης θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να συντάξουμε μια χρήσιμη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που θα τονίσει τη σημασία του εμπορίου με το Ιράν μετά την υπογραφή της πυρηνικής συμφωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά, συζητάμε ταυτόχρονα και το σημείο 8, δηλαδή τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα ήθελα λοιπόν να πω κάτι πάνω σε αυτό, εκ μέρους της κυρίας Χάκε. Μετά την υπογραφή λοιπόν της συμφωνίας αυτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεσμεύτηκαν να ανούν όλες τις κυρώσει Όμως οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβλήματα στις ε, συναλλαγές τους ε, με το Ιράν εξαιτία των Αμερικανικών κυρώσεων που δεν έχουν ακόμα έρθει. Αυτή η εξοεδαφική ε, επιρροή έχει λοιπόν επηρεάσει αρνητικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε με προφορική ερώτηση να απαντηθεί το τι έχει γίνει για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν περισσότερη ασφάλεια δικαίου και ένα φιλικότερο περιβάλλον στις συναλλαγές τους με το Ιράν. Σκοπεύουμε να ε, συζητήσουμε το θέμα αυτό αύριο και να ε, το πάμε στην Ολομέλεια το συντομότερο δυνατόν. Με χαρά μας λοιπόν θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. 25 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών, 6 το απόγευμα. Και πράγματι η προφορική αυτή ερώτηση θα εξεταστεί αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν και το τελευταίο σημείο της ε, ανοιχτής συνεδρίασης. Θα συνεχίσουμε με την συνεδρία των συντονιστών.